Maman. Start. We come to the human rights, democracy. Ξεκινάμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία. Ο κύριος Λάμστορφ είναι ο εισηγητής. Σωστά. Πού είναι. Άντρου θα αναλάβεις εσύ γιατί εκείνος είναι στη Λιβύη. Θέλεις να πεις κάτι? Όχι. Μια που δεν είναι ο Χραφ Λάμστορφ μαζί μας σήμερα, γιατί είναι στη Λιβύη, έχει εκεί αναλάβει καθήκοντα για την πρόθεση της δημοκρατίας, πάντα χρειάζεται. Ας αρχίσουμε Τροπολογία 93. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Να αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. 23 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Γυναικών 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε έτσι φτάνουμε στην τροπολογία γυναικών 8, φεμ 8. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες. 21 ψήφοι υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές. 103 ξανά παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Πέρα στις ψηφοφορίες. Κυρία Κράτσα, δεν έχετε τύχει σήμερα. 27-25 απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες. 30 υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά αποχές δεν είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα στις φοφοριες 29 29-19 εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά Ας ελέγξουμε καλύτερα. Πέρας της ψηφοφορίας. «25-25 είναι το αποτέλεσμα, απορρίπτεται». Τώρα είμαστε στην 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165. Να, όχι, καταπίπτει αυτή. Φεμ 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17, 124 και 125 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 126 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 127-128, α, καταπίπτει αυτή, οπότε φτάνουμε στη 18 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ερχόμαστε στην 20. Κατά αποχές δεκτή. 33 και 134 αποχές δεκτή. 12 γυναίκες υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 γυναίκες έχει εκπέσει 13 ε, γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 γυναικών υπέρ. Κατά. Δεκτή. 15 γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Δεκτή. 130. 6 εκπίπτει. 137 υπέρ. 137 υπέρ. Υπέρ. Κατά από... Πάλι, πάλι. Υπέρ. 137. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 138. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο 139. Είπαμε ότι απορρίφθηκε. Δεν κατάλαβα τους σοσιαλιστές ποτέ. Λέει ο πρόεδρος. Πέρας ψηφοφορίας, εν πάση περιπτώσει. Δεν το, δεν το ζήτησα εγώ. Ποιος, ποιος, ποιος ζήτησε έλεγχο. Παίρνουμε με κέρας μια μπύρα. Κάποιος από εδώ. 16 γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18 γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σκάνουμε. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή, αλλά κάνουμε έλεγχο, λέει ο πρόεδρο. Πέρασε ψηφοφορία. 29-21 γίνεται δεκτή. 17 ε, ντεβε υπέρ, κατά, αποχέ απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά, Αποχέ, απορρίπτεται. 143 και 144 υπέρ κατά αποχές δεκτές. ΔΕΒ 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Απορρίπτεται, απορρίπτεται, συγγνώμη. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΔΕΒΕ 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται γυναικών 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. 151 υπέρ κατά αποχές δεκτή 152 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή Πάμε στην 158 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒ 23 υπέρ κατά δεκτή. ΔΕΒ 24 έχει εκπέσει 24. Μα αυτή ψηφίσαμε τώρα. Όχι την 23. Φέμ 20, 20 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. «164 υπέρ» κατά αποχές δεκτή. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φέμ 21 υπέρ κατά. Δεκτή. Έλεγχος, βεβαίως, έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 168 έχει εκπέσει, 169 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒ 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΦΕΜ 23. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 28 υπέρ. Θέλετε έλεγχο στη ΦΕΜ 23. Άρχεται η ψηφοφορία έλεγχο. Ναι. Δεκ... Συγγνώμη. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Έχει εγκριθεί. 28 ψήφι υπέρ κατά. Αποχές δεκτή. 10 προϋπολογισμών υπέρ κατά. Αποχές δεκτή. 171 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Φέμ 24 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 του εισηγητή υπέρ κατά. Αποχές δεκτή. 30 υπέρ κατά α, απο, γίνεται δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 182 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35, 36, 37, 35, 36, 37 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέμενα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θεμ 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή. 40 με προφορική τροπολογία 2 ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. ΔΒ1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. ΦΕΜ 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά 45 υπέρ κατά δεκτή 46 υπέρ Σαράντα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά κάνουμε έλεγχο. Πέρασε. Γίνεται δεκτή 27-23. Φεμ 4. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΔΒ3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 προϋπολογισμών υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Φεμ 6 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 13 <clears throat> υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προϋπολογισμοί 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 14 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 8 προπολογισμών εκπίπτει. 92 εκπίπτει. Εντολή διαπραγματεύσεων. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Πω, Θα γίνω στουπί στο τέλος αυτής της συνεδρίασης, λέει ο πρόεδρος. 49, 0 κατά και 4 αποχές. Πρέπει να το αναφέρουμε στον κύριο Λάμψο, τον πάρουμε τηλέφωνο στη Λιβύη. Τώρα ερχόμαστε στην έκθεση της κυρίας Γκόμες, η οποία όμως δεν είναι εδώ. Ίσως ακολουθεί κατά πόδα στον κύριο Λάμστορφ στην Λιβύη, η κυρία Γκόμες. Ποιος εκπροσωπεί την κυρία Γκόμες? Κυρία Μουνής, μάλιστα. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 11. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 52 υπέρ κατά Πρέπει να ελέγξουμε. Έλεγχο στην 52. Πέρασε. 26-25. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρι... Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. 22-23 απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63, 64, 65 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτές. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες Μπραντνερ μέχρι την 71. Υπέρ, κατά, απόχες, δεκτές. 72. Υπέρ, κατά, απόχες, δεκτή. Προφορική 2. Υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τις υπόλοιπες τροπολογίες Μπράντρε μέχρι την 30... Όχι, μία-μία. Δύο την ψηφίσαμε υπέρ. Το κάναμε. Έχει εγκριθεί. 31. Ο κ. Μάουρο θέλει να πει κάτι. Πρόκειται για μια προφορική τροπολογία, την οποία έχω ήδη προτείνει στην εισηγήτρια και είναι υπέρ. Θα σας το διαβάσω στην αγγλική γλώσσα. Για την αναπτυξιακή πολιτική αυτό που έχει σημασία είναι οι εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ε, παρεμποδίζουν τις προσπάθειες των τρίτων χωρών σχετικά με το άρθρο 208 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνείτε κυρία Μπράντνερ. Ναι, η κυρία Μπράντνερ δέχεται αυτή την ε, τροποποίηση. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 33 <clears throat> υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 37 υπέρ κατά αποχές ε, έλεγχος για την 37. στις πληροφορίε. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές Έλεγχο. Πέρας. Απορρίπτεται 26-28. 5 του εισηγητή υπέρ της κατά αποχές 6 της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το σύνολο με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πραγματικά συντριπτικά. Συντριπτική πλειοψηφία. Παγκόσμιο ρεκόρ. Θέλετε έλεγχο. 54 συν καμία ψηφοσκατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην απούσα εισηγητρία η οποία διάλεξε το σωστό δρόμο και δεν ήταν στη συνεδρίασή μας, την κυρία Γκόμπης. Τώρα, ερχόμαστε στην έκθεση Μπραντνερ το μέσο σταθερότητος. Κύριε Μπραντνερ, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 92 υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 94 υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 96 Συγγνώμη, συγγνώμη, DV5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 96 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην... 13 ε, ψήφι υπέρ κατά, αποχές δεκτή, DV7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 100 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 101 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 102 υπέρ, κατά αποχές δεκτή συμβαστική 6 <clears throat> παρακαλώ θέλετε έλεγχο στην 102 102 μάλιστα Εκατόν δύο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 35-18. Δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 106 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 7 προϋπολογισμών, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Check, check. Έλεγχος. Περισσεύουν κάποιοι πράσινοι εδώ. Και χθε είχαμε 7, έτσι δεν είναι. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Πέρασε ψηφοφορία. 30 με 25 δεκτή. Ήταν η προπολογισμού 7. 17 υπέρ κατά άποχες δεκτή 109 υπέρ μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογιες λεζινγκ Λόζινγκ από κοινού 109-123 υπέρ κατά άποχες απερίφθησαν προϋπολογισμός 8 υπέρ κατά άποχες δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προπολογισμών 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 127 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές DV10 υπέρ κατά αποχές δε... 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 130 υπέρ 31 συγγνώμη κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμών 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Θέλετε έλεγχο. Έλεγχος στην 11 προϋπολογισμών. Πέρας ψηφοφορίας. Απέριπτε. 23-30. Απέριπτε. 28 υπέρ κατά αποχές η ίδια πλειοψηφία. Έλεγχος. Πέρασε. 13.40. Ακόμα καλύτερα. Απορρίπτεται αρχίζει να εμφανίζεται μια σιωπηρή πλειοψηφία η οποία δεν είχε συμμετάσχει προηγουμένως. Λέω πρόεδρος. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος για την 30. Πέρας. 26-25 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 33 υπέρ αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 146 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά <clears throat> αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 153 υπέρ κατά έλεγχος. Πέρας. 32-24 δεκτή. 44 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 46 με την προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 154. Όχι, όχι, όχι, έχει εκπέσει. 47 DV20 υπέρ κατά αποχές. 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μάλλον απορρίπτεται, συγγνώμη, απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ίντε 2 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. τα 3 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Είναι τα 3. Πέρα τη ψηφοφορίες. 26 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. περίπου πέρας της ψηφοφορίας, πέρας τώρα της ψηφοφορίας, απορρίπτεται 27-27 είναι το αποτέλεσμα. ΔΕΒ 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ίντα 4 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 26-30. Απορρίπτεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 167 υπέρ, 166 πρόεδρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύε 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα υπέρ, α 171 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 100... 72 ξανά υπέρ, κατά, αποχές. Ναι, έπρεπε να το έχω καταλάβει. 173 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε καλύτερα. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Πέρα στις φοφορίες. 22-32 απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 178. Μπορούμε να ψηφίσουμε 178 με 186 μαζί, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. 61. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ίντε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 64 κατά πίπτη, 64 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι 8 κατά πίπτη, 65. Εδώ έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία. Κύριε Μπράτνερ, μπορείτε να μας το εξηγήσετε παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω απλώς να προτείνω κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο, να δώσει κατάλληλη απάντηση στα θέματα δημόσιας υγείας όσον αφορά διάφορες επιδημίες αυτό να μείνει και να καταψηφίσουμε το σχέδιο ε, πήγουσας ανάγκης και τα λοιπά να εξαιρεθεί από το κείμενο. Ευχαριστώ. 65 υπέρ. Πρώτο τμήμα. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΔΕΒ 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΔΒ3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 94 κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 6 σε τρία τμήματα η έξι. Υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, θα ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα. Πέρα στις ψηφοφορίες. 29-27 εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κύριε Μπρότνερ, βλέπετε 85 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά. Οι σοσιαλιστές ψηφίζουν υπέρ ή όχι. Α, κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 89 υπέρ. 10 μάλλον τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογισμή 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογισμή 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογισμή 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα για τη διαπραγματευτική ε, εντολή ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 54 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά και καμία αποχή. Κύριε Μπράντνερ, Ευχαριστώ τους και εισηγητές, τους οφείλω πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Μάρκος, ο οποίος θα επιστρέψει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας σύντομα, αλλά έκανε μια εξαιρετική δουλειά εδώ στη γραμματεία της Επιτροπής μας. Κυρίες και κύριοι, πριν αλλάξουμε εδώ στο Προεδρείο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κέλλα, με έχει γενέθλια σήμερα. So colleagues, we have uh, still... You want to do it from there? Oh, I can, I can, okay. Αναλαμβάνω εγώ, λέει ο κύριος colleagues, we can uh, Ξεκινάμε με την τελευταία ψηφοφορία. Πριν από τις... Ε, όχι, δεν είναι η τελευταία, λέει ο κύριο Μπρόκ. Α, δεν είναι η τελευταία, <laughs> έχουμε κι άλλε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την DEV ε, 16. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εποχέ δεκτή. Είναι τα δύο υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. ΔΕΒ 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 3 και ΔΕΒΕ 18 ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Α, έχει καταπέσει η 39. Συγγνώμη, για μια στιγμή λέει ο πρόεδρος. Α, θα ψηφίσουμε 39 τελικά υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μετά περνάμε στη συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δώδεκα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεκατρία υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 43 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεκατέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ήταν ταυτόσημη με την ΤΕΒΕ e 26, περνάμε στη 45 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΔΕΒΕ 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε στην Δεύε 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύε 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Deve 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Deve 32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Budget 14 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Deve 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή Δεύε 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Budget όχι για μια στιγμή λέει ο πρόεδρος Budget 15 ναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πρέπει να ψηφίσουμε και την 54 λέει ο πρόεδρος. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 και 56 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ντεβε 35 και Ίντα 7 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύε 36 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 59 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 61 παρακαλώ ψηφίζεται. Please close the vote. ψηφοφορίας. Την 61. Έγινε δεκτή. Δύο ταυτόσημες, οι 62 και 63 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Τροπολογία 65 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 19 ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ντεβε 40 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 67 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Είναι τα 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δέβε 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. budget 17 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην 73. Α, για μια στιγμή. Εδώ μας λείπει η διατύπωση. Κύριε Μπρόκ έχετε το λόγο. Μετά από πρόταση της κυρίας Μπράτνερ έχουμε μια νέα διατύπωση αλλά σε πιο ξεκάθαρη γλώσσα. Θα πρέπει να δίδονται ε, αυτά τα ποσά στο Ταμείο για την Πρόθωση της Δημοκρατίας έτσι ώστε οι χώρες αυτές να μπορούν να ε, τις ενισχύσουν. Και όταν τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να δοθούν λόγω των ε, ε, δύσκολων τοπικών συνθήκων, τότε θα τροφοδοτούν το Ταμείο αυτό για τη Δημοκρατία. Αυτή είναι η νέα σας διατύπωση της τροπολογίας 73. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της νέας διατύπωσης. Κατά. Αποχές. Θέλετε το λόγο κύριε Τάνοκ, κάτι είπε ο κύριος Τάνοκ εκτός μικροφώνου. Ε, ο κύριος Μπρόκ είναι εισηγητής και είχε μια προφορική τροπολογία, λέει ο κύριος Κόβατσεφ. Κύριος Τάνοκ συνέχισε εκτός μικροφώνου. Δεν κατανοώ τις παρατηρήσεις σας, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ψηφίζουμε την 73 με την προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Πηγαίνουμε στην 19 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Budget 21 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 74 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 75 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 76 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Κυρία Μπραντνερ έχετε το λόγο σύντομα πρόεδρε η τροπολογία αυτή θα πρέπει να προηγηθεί τις 77 αλλά η ουσία δεν αλλάζει απλά η θέση Η 79 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 80 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 και 83 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Αδεκτές ΔΕΒΕ 45 και ΔΕΒΕ 46 υπέρ, κατά, αποχές, δε, απορρίπτονται. Είναι τα 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 48 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε τώρα στην 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ψηφίζουμε ομαδών την budget 22 και 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 20 αποσύρεται. 89 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε την 90 υπέρ. Όχι, έχει καταπέσει λέει ο κύριος Μπρόκ η 90. Πρέπει να ψηφίσουμε τώρα την 90 όμως επιμένει ο Πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 90 και ντεβε 50 από κοινού. Πέρα στις ψηφοφορίες. δεκτή 26 υπέρ 24 κατά. Περνάμε τώρα στην ΤΕΒΕ 51 υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την ΤΕΒΕ 51. Απερίφθη. Ίντερ 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Πηγαίνουμε στην ΤΕΒΕ 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22 ψηφίζεται. Πέραση ψηφοφορίας. Δεκτή. Λοιπόν, 98 και ντεβε 54 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Ντεβε 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ντεβε 56 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 100 και budget 29 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Είναι τα 18 και 19 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Budget 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Dev 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Dev 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Dev 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Περνάμε τώρα στην 26 υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο ηλεκτρονική ψήφος για την 26. Απορρίπτεται 27 κατά και 25 υπέρ. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 και budget 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. ΔΕΒΕ 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Budget 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στη συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην 8 του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 9. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προϋπολογισμός 9. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 38. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές. Η 38 ηλεκτρονικά ψηφίζεται αν και νομίζω ότι απερίφθη. Ψηφίζουμε την 38 ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 26 ψήφοι κατά. Προϋπολογισμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συνεπώς τώρα έχουμε την, την εντολή, ηλεκτρονική ψήφος για την εντολή. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. «49 υπέρ κανείς κατά τρεις αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Μπροκ». Yeah. I was too optimistic, I forgot the last. Ήμουνα πολύ αισιόδοξο. Είχα ξεχάσει ότι έχουμε άλλη μια ψηφοφορία. Μια τελευταία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Ευθύσαμε στους 28 τροπολογία υπέρ. Ναι, γυμναστική, κύριε Κασουλίδη, είναι καλό για την υγεία. Γυμναστική. Τροπολογία 28, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, συνάδελφοι, πρέπει να ψηφίσουμε την 30 πρώτα απ' όλα του κ. Πάσκου υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμβαστική 30 εγκρίνεται. Η τροπολογία 30 διορθώνω πρόεδρο. Συμβαστική 1 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Κατά τμήματα. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Τη 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Για τη 48 λοιπόν θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άλλοι 7 πρέπει να ψηφίσουμε. Άλλοι 6, 5... Πέρα στις ψηφοφορίας. Με μία ψήφο απορρίπτεται. Συμβαστική δύο υπέρ. Συμβιβαστική δύο. Ένα πρόβλημα με το ΕΛΚ υπάρχει. Δεν ψηφίζουν. Περίεργο. Θα πρέπει να ήταν ε, σύνεδο. εδώ. Δύο. Υπέρ, παρακαλώ, τη συμβαστική δύο. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. 56 διορθώνω ο πρόεδρος. Πρέπει να ψηφίσουμε την 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 59. Ωραία. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται με 27 ψήφους κατά και 21 ψήφους υπέρ. 60 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε για την 72 παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία κατά. 73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 84. Ωραία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άλλοι πέντε πρέπει να ψηφίσουν. Έχουν τις κάρτες τους στο μηχάνημα, αλλά δεν ψηφίζουν. Πέρα στις ψηφοφορίες τώρα. Απορρίπτεται. Με 28 ψήφους κατά, 21 ψήφους υπέρ. 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89 ε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 κατά τμήματα, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 101 παρακαλώ. Πέντε λείπουν ακόμα, πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται, 25 ψήφι κατά. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120 με προφορική τροποποίηση. Ψηφίζουμε με την τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 122 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα Τη 122. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται πράγματι με διαφορά δύο ψήφους και μία αποχή. Τώρα, συμβαστική 6. Υπάρχει προφορική τροποποίηση του εισηγητού. Παρακαλώ κύριε Μπρόκ. Υπάρχει μια συμφωνία νομίζω μεταξύ ΕΛΚ και σοσιαλιστών τουλάχιστον, ίσως κι άλλο, να δείτε το κείμενο της συμβαστικής 7. Σημείο 6 που μιλάει για την πόλωση όσον αφορά την τουρκική κοινωνία, τώρα πρέπει να λέει ότι η εμβαθυνόμενη πόλωση στην τουρκική κοινωνία. Θα έλεγα να ψηφίσουμε το συμβασμό με αυτόν τον τρόπο και να συμφωνήσουν όλοι όσοι συμφώνησαν και με τη συμβαστική. Ο κύριος Νταφ, εγώ δεν βλέπω τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Κύριε Νταφ, θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Νταφ. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν αναφερόμαστε μονάχα στον διχασμό μεταξύ κοσμικών και θρησκευωμένων, αλλά μιλάμε γενικά για την πόλωση στην ε, τουρκική κοινωνία, ότι περιλαμβάνει το στοιχείο αυτό της θρησκευτική διαίρεσης, αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο πόλωση. Μιλάμε γενικά για την αυξανόμενη πόλωση στην τουρκική κοινωνία, χωρίς να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το θέμα της κοσμικότητας, της εκοσμίκευσης ή της θρησκείας. Κύριε Ντάφ, αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνούμε για αυτό το θέμα, τη συμβαστική αυτή τροπολογία 6 με την προφορική τροποποίηση του εισηγητού βεβαίω. Εντάξει, ψηφίζουμε. Συμβαστική 6 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με την προφορική αυτή τροποποίηση. 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή 128 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται οι τέσσερις τροπολογίες του κυρίου Μάιερ από κοινού 130, 131, 132, οι τρεις αυτές τροπολογίες από κοινού του κύριου Μάιερ. Όχι, δεν θέλετε μαζί. 130, μόνη της, υπέρ. Την έχουμε ψηφίσει την 129. Υπήρξε διπλή εγγραφή στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ο δαίμον του τυπογραφείου. Ψηφίσαμε την 129 λοιπόν. 130 υπέρ. Κατά. Απόφε, αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές 144 υπέρ κατά <coughs> χρειάζεται έλεγχος 144 ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ Πέρας. Εγκρίνεται. 23-20. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για 147. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20-27, 148 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά συ... καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία. Γιατί έχει γίνει δεκτή η τροπολογία 6. διαφορετικά πράγματα λένε οι κατάλογοι ψηφοφορίας μας. Ο εισηγητής. Εφόσον έχουμε δεχτεί την τροπολογία 6 είπαμε ότι καλύπτει όλες τις τουρκικές τροπολογίες, λέει ο κύριος Μπροκ. Νομίζω ότι υπήρχε ένας παλιός κατάλογος και είχε διανεμηθεί ένας νέος κατάλογος. Είπαμε όλα αυτά τα οποία λέγονται στην Τουρκία καλύπτονται από τη συμβαστική τροπολογία 6. Σας παρακαλώ να δεχτείτε λοιπόν αυτή τη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ των σκιωδών εισηγητών χθε το βράδυ. Όλα τα θέματα μέχρι το 69α καλύπτονται από την τροπολογία 6, τη συμβαστική. Ας ακολουθήσουμε αυτά που λέει ο συγητής μας. 166. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται 167. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 168. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 169. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 170 <clears throat> με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ πάλι προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές ασαφές πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 172 άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται 21-25. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δεύτερο τμήμα του 879, ηλεκτρονικό έλεγχο, εγώ νομίζω ότι απορρίπτεται. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Όχι δικιά μου, λέει ο κύριο Μπρόκ. 180. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές δεκτή 186 υπέρ κατά αποχές δεκτή 187 υπέρ σε δύο τμήματα μάλλον πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Που είπαν ότι το δεύτερο τμήμα εκπίπτει διότι έχουμε εγκρίνει τροπολογία 181. «187 δεν την ψηφίζουμε διότι εκπίπτει, συγγνώμη, 188 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος για την 188. Πέρας. Εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 191 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 191. Κυρία Λούνατσεκ, έχετε το λόγο να λάβω το λόγο για την 191 ως σκιώδης εισηγήτρια. Θέλω να ζητήσω από τον κύριο Λίζεκ να αποσύρει την προφορική του τροποποίηση γιατί δεν είχε τύχη συμφωνίας μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και ζητώ από όλους να καταψηφίσετε αυτή την τροπολογία γιατί στις συμφωνίες σύνδεσης που ψηφίσαμε την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν είχαμε μια διαφορετική διατύπωση και θέλω να αναφερθώ σε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν μιλήσουμε για περιοχές όπως η Απχαζία σαν κατεχόμενα εδάφη και όχι στον Αγκόνο Καραμπάχ ως κατεχόμενο έδαφος, αυτό είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και δεν πρέπει τώρα να το κάνουμε σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί στρέφεται εναντίον των δύο άλλων συμφωνιών σύνδεση που ψήφισαμε σε αυτό το κοινοβούλιο. Ζητώ πρώτα τον κύριο Λίζεκ να πω. Σύρει την προφορική τροπολογία για την ελληνική συμφωνία μεταξύ των σκιωδών και επίσης ζητώ από όλους να καταψηφίσουν για τους λόγους που ανέφερα δύο μέτρων και δύο σταθμών. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Από τη σοσιαλιστική ομάδα εμείς συμφωνούμε απόλυτα με την κυρία Λούνατσικ. Λαντσπέργκης. Σας ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Η τροπολογία αυτή, χωρίς, μικρό... χωρίς μικρόφωνο, κύριος Λαντσπέργης, Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται ο κύριος Ζαντσπέργης. Κύριε Λανσπέργης, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Τώρα ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε υπέρ ή όχι κατά. Μα Όλα αυτά που λέγονται για τον Αγκόνο Καραμπάχ είναι πραγματικότητα, λέει ο κ. Λαντσμπέργκη, χωρί μικρόφωνο. Μα δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Μόνο στον εισηγητή μπορώ να δώσω το λόγο και μετά θα ψηφίσουμε. Παρακαλώ, ο εισηγητή, κ. Μπλοκ. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια συμβαστική λύση. Αν πάρετε το αρχικό κείμενο και παραμείνουμε σε αυτό. Αλλά να περιλάβουμε το θέμα της ε, κατοχής από τη Ρωσία της Νότιας Οσετίας και της Απχαζίας. Να κρατήσουμε το κείμενο όπως είναι, αλλά να μιλήσουμε και για την Νότια Οσετία και την Απχαζία. Γιατί αν μιλήσουμε μόνο για τον Αγκόνο Καραμπάχ και την υπερνηστερία και δεν μιλήσουμε για τη ρωσική κατοχή της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας, αυτό είναι διπλωμέτρα και δύο σταθμά. Εντάξει, αν δεν το δέχεστε αυτό, ας ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία του κυρίου Λίζεκ. Συνάδελφοι, δεν μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε συζήτηση. Μα δεν είναι συζήτηση, λέει η κυρία Κοπά. Σοσιαλιστική ομάδα. Επειδή είναι μια προφορική τροπολογία, ακόμα και αν ένα μέλος αντιταχθεί, δεν μπορεί να ψηφιστεί. Ναι, εγώ, την, ε, εγώ αντιτίθεμαι, λέει κύριε Κοπά. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία. Είναι πολύ απλό. Ψηφίζουμε λοιπόν την, την 191, 191 χωρίς την προφορική τροποποίηση. 191 ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 191. Πέρας. Απορρίπτεται. 22-26. Δεν γίνεται δεκτή η τροπολογία 191. 1-9-2. <clears throat> Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 193. Πέρας. 29-18 γίνεται δεκτή. Τροπολογία 194 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Θέλετε να κάνετε έλεγχο. Έλεγχος για την 194. Πέρας. Απορρίπτεται 20-27, 196 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...212 με προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 2.13 του κ. Σφόμποντα. Πέρας εγκρίνεται 2.18 υπέρ κατά αποχές πάλι πρέπει να ελέγξουμε για τη 218 πέρας εγκρίνεται 2.21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.23 με προφορική τροπολογία κατά αποχές εγκρίνεται. 2.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 226 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 227 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 228 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 229 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 230 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 231 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 235 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε καλύτερα. 236. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 237 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 238 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 239 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 230 υπέρ, 240 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 242 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. 242 πρώτο τμήμα. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εδώ Μένουμε όλο και λιγότεροι. Απορρίπτεται 21 ψήφοι κατά και 18 υπέρ. Δεύτερο τμήμα τώρα τη 242 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο. Απορρίπτεται. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 244. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 246 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 247 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 248. 247 αν θέλετε. Ωραία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. 248 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 249 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 250 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 251 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 252 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. 253. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέσσερις δεν ψηφίζουν. πέρες ψηφοφορίας εγκρίνεται 26-19. 254 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 258 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 265 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 266 υπέρ, κατά, πρέπει να ελέγξουμε. 266 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ, 20 κατά. Τροπολογία 267, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 268 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 269 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 269. Δεν ήταν πολύ σαφέ το αποτέλεσμα. Ψηφίστε παρακαλώ. 269 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Τώρα, τροπολογία 270. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 271 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 271. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. 272 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 273 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 273 απορρίπτεται λέω εγώ, αλλά αν θέλετε θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Άλλοι τέσσερις μένα να ψηφίσουν. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 20 κατά, 18 υπέρ. 274 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 276 με προφορική τροπολογία υπέρ. Προφορική τροπολογία ή 11 είναι η προφορική τροπολογία. Παρακαλώ κυρία Μουνής. Ευχαριστώ. Έχουμε έναν κατάλογο ψηφοφορίας που πήραμε 15 λεπτά πριν την ψηφοφορία. Δεν είχαμε την ευκαιρία να ελέγξουμε τις προφορικές τροπολογίες. Παρακαλώ τότε τον εισηγητή διαβάσει. Περιλαμβάνει δύο λέξεις μόνο. Ότι ο συμβασμός βασίζεται στο δίκαιο και ελεύθερο εμπόριο. Όχι μόνο δηλαδή θεμητό εμπόριο. και στηρίζει βασικά την τροπολογία σας. Συμφωνούμε με την προφορική αυτή τροπολογία. Ωραία, ψηφίζουμε. Τότε 276 με την προφορική αυτή τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 277 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 278, πάλι με προφορική τροπολογία, αριθμός 12. Υπέρ, θέλετε να την ε, διαβάσουμε. Να τη διαβάσει ο εισηγητής την ε, προφορική τροπολογία αριθμός 12 δηλαδή. Ναι, λέει στο τέλος δεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ασχοληθεί με όλες τις συμφωνίες για την Αφρική προκειμένου αυτές να, είναι, να ενισχύουν την αποτελεσματική πολιτική. Ε, βασικά χρησιμοποιεί το συμπέρασμα της δικιάς σας τροπολογία κύριε Μπράτνερ. Θέλετε το λόγο κύριε Μπράτνερ. Όχι. Πρόεδρος. Αν συμφωνούμε λοιπόν για αυτή την προφορική τροπολογία, ψηφίζουμε υπέρ τη 278 κατά αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 278 με προφορική τροπολογία. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 22-22. Άρα ψηφίζουμε τη 279. Η 278 μόλις απορρίφθηκε με ισοψηφία. Τώρα 279 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 280 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 280. Πέρα στις φοφοριες εγκρινεται Εγκρίνεται. 24-19. 282 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 283 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 284 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 285 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της 285 παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 286 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 287 υπέρ. ...287. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Αλλά να ελέγξουμε. Έξι συνάδελφοι με να ψηφίσουν ακόμα. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 288 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 289 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ και αυτήν. 289. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται 23 υπέρ 20 κατά. 290 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 291 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 292 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. 292, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε τις εγκρίνεται. 293 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 294 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Α, κυρία Μπράντνερ, παρακαλώ κύριε Μπράτνερ. Σας ευχαριστώ για την επόμενη αυτή τη συμβαστική 10 υπάρχει κατά τμήματα ψηφοφορία που έχουμε ζητήσει, αλλά εδώ αναφέρεται λάθος, δεν είναι όπως το θέλαμε. Το πρώτο τμήμα πρέπει να πηγαίνει μέχρι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και για τα δύο... Θέλουμε να πούμε ότι και τα δύο τμήματα πρέπει να καταλήξουν σε μια συμφωνία όσον αφορά την εμπορική συμφωνία με την Ινδία υπέρ του δίκαιου εμπορίου και της ανάπτυξης. Σε αυτό το τμήμα είναι που θέλουμε εμείς την κατατμήματα ψηφοφορία. Για επαναλάβετε παρακαλώ που θέλετε να χωριστεί. Συγγνώμη αν υπάρχει σύγχυση. Το έστειλα σωστά, αλλά κάπου χάθηκε. Και για τα δύο τμήματα να καταλήξουν τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη διάσκεψη για την εμπορική συμφωνία με την Ινδία, η οποία θα ενισχύσει το εμπόριο και την ανάπτυξη. Αυτό θέλουμε χωριστά ξεκινάει και τα δύο τμήματα και πάει μέχρι την οικονομική ανάπτυξη. Το άλλο μένει εκεί. Λοιπόν, χωρίς αυτή την πρόταση ψηφίζουμε πρώτα και μετά θα ψηφίσουμε αυτή την πρόταση. Συνεπώς, πρώτο τμήμα, χωρίς δηλαδή αυτό το τμήμα που μόλις μας διάβασε η τρίπερ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα, αυτή την πρόταση ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 304 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 305 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. 305. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. Λοιπόν, εκκρίνεται με διαφορά μία ψήφο. 306 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 307 υπέρ. Αφού απορρίφθηκε 306. 307 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 308 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «313 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 317 τώρα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 318 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 319 υπέρ, κατά, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 319 ψηφίστε. Πέρας της φοφορίες. Απορρίπτεται. 19-25. 320. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 321 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 322 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 323 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 324 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 325 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 326-327 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 328 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 329 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 330, όχι, 330 ναι, ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 331. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατά. Αποχές. Αυτό θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Το δεύτερο τμήμα, το τρίτο τμήμα μάλλον, κατά, αποχές, δεκτή. 3.32 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3.33 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3.34 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3.35 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 3.36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.37 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3.38 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3.39 υπέρ. Κατά. Πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος στην 3.39. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πηγαίνουμε τώρα στην 3.40 και 3.41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. ...3.39 έχει γίνει δεκτή, έχει απορριφθεί, συγγνώμη. Ψηφίζουμε τώρα την 3.42. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 343 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 344 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 345 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 347 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 348 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 349 υπέρ κατά Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 349. Πέρα της ψηφοφορίας. Ο εισηγητής θα ήθελε το λόγο. Μια άλλη τροπολογία η οποία συνδέεται έχει απορριφθεί, δεν έχει πλέον νόημα το κείμενο, είναι θέμα σειράς. Αν απορριφθεί ο τίτλος δεν μπορεί να αλλάξει ο επόμενος. Δεν θα πρέπει να την ψηφίσουμε και θα κάνω εγώ εκ των υστέρων μια πρόταση στην Ολομέλεια για να λυθεί το θέμα που δημιουργείται. Μην ψηφίζουμε λοιπόν. Ακολουθούμε. Α, η κυρία Μονής έχει δει το λόγο. Μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα εγκρίνουμε με την προφορική τροπολογία. Γιατί αν η συγκεκριμένη τροπολογία δεν έχει νόημα δεν έπρεπε να κατέβει για ψηφοφορία. Και όχι να λέμε εκ των υστέρων ότι δεν τίθεται θέμα ψηφοφορίας. Μπούτι κόφερ. Κοιτάξτε, εμείς ψηφίσαμε ό,τι ψηφίσαμε, αλλά παρόλα αυτά η προφορική τροπολογία θα κατατεθεί στην Ολομέλεια. Αυτό λέω και εγώ, λέει ο κύριος Μπρόκ. Κοιτάξτε, η 349 δεν έγινε δεξή. Μα την καταψηφίσαμε την 349, οπότε δεν έχει νόημα το κείμενο. Λόγω ακριβώς της κατάστασης που δημιουργήθηκε να μου επιτρέψετε μαζί με τον κύριο Πάσκο να καταθέσω μια συμβιβαστική ή μάλλον μια προφορική στην Ολομέλεια. Το πρώτο τμήμα απερίφθη, οπότε το να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, ας ακολουθήσουμε τη σύσταση του εισηγητή. Μαζί με τον κύριο Πάσκου θα κάνουν πρόταση στην Ολομέλεια. Περνάμε στην 352. Το ίδιο θέμα τίθεται και με το 352. Δεν είναι θέμα περιεχομένου, είναι θέμα τάξης, θέμα σειράς. Σας έχουμε εμπιστοσύνη λοιπόν. Η 351 είναι η επόμενη, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 352 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 353 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 3.55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.58 με προφορική τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε στην 363. Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή 364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 365 και 366 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 367 υπέρ κατά αποχές δεκτή 368 υπέρ κατά αποχές δεκτή 369 υπέρ κατά δεκτή 370 υπέρ κατά αποχές δεκτή 371 υπέρ κατά αποχές δεκτή 372 υπέρ κατά αποχές δεκτή 373 υπέρ κατά αποχές δεκτή 374 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 375 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 376 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 377 υπέρ κατά αποχές δεκτή 378 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 378 παρακαλώ. Απορρίφθη. Απερίφθη, συγγνώμη. Προσπάθησα και Βανόρντεν όπως είδατε. 3,79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3,80 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 381 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 12 υπέρ Κοιτάξτε υπάρχει ένα λάθος λέει ο, ο πρόεδρος ο κύριος Μπροκ. Υπέρ. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ναι λέει ο κύριος Μπροκ. Η γραμματεία μας εδώ έχει κάνει λάθος. Κατά. Αποχές. Η συμβιβαστική 12 γίνεται δεκτή. 389 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 390 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 391 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 392 υπέρ κατά αποχές δεκτή 393 υπέρ κατά αποχές δεκτή 394 υπέρ κατά αποχές δεκτή 395 υπέρ κατά αποχές δεκτή 396 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 396. 3.96 λοιπόν. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη με μία ψήφο. 3.96 λοιπόν απερίφθη. Η 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Η 7 υπέρ. Η 7 υπέρ λέγω κατά αποχές δεκτή. Η 8 Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον κατάλογο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τις 7 και τις 8. Με την 8 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Η 12 μαζί με την προφορική 15. Αν θέλετε να την πούμε προφορική 13 γιατί όχι. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 και 16 είναι ταυτόσιμες κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 αλλά και 22 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 23 υπέρ κατά πρέπει να κάνουμε έλεγχο στην 23 ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 17-24, τροπολογία 24 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 με προφορική τροποποίηση 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 27 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές για την 27, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5 βεβαίως απορριπτεται Απορρίπτεται. 18-23. Τώρα, τροπολογίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Προϋπολογισμοί 2 υπέρ. Υπέρ. Η ένα καλύπτεται, η δύο δεν καλύπτεται, είναι ακάλυπτη. Δύο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα προϋπολογισμών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Budget 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ηλεκτρονικά για το σύνολο της έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί άρχεται. Ψήφισατε όλοι και όλες. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Ήταν η πιο σημαντική μας έκθεση. 34 ψήφοι υπέρ, μία κατά, 6 τροπολογίες. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπρόκ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία που έδειξαν, τους σκιώδεις εισηγητές. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι αναπόφευκτο, να μην είναι απόλυτα σαφή και να μην έχουν διευκρινιστεί, θα πρέπει να προετοιμαστούμε στην Ολομέλεια να έχουμε επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπροκ. Η κυρία Λέζιν θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι εμείς εξ ονομάτων της ομάδας της ΓΚΟΕ θα υποβάλουμε μια έκθεση μειοψηφία. Εντάξει. Η γραμματεία θα το καταγράψει. Σας ευχαριστώ για την, για την ε, υπομονή σας και σε λίγα λεπτά θα συνεχίσουμε με την ημερησία διάταξή μας. Σημείο 16 ημερήσιας διάταξης τώρα. Έκθεση Μπραντνα για την διαθεσμική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιών σε σχέση με τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και για την υγεία δημοσιονομική διαχείριση. είναι σημαντικό το τελευταίο στοιχείο, το Sound Financial Management. Έχετε το λόγο κυρία Μπράντον, σας ευχαριστώ. Είναι θέμα χρημάτων. Πολλοί από εσά είσαστε, για εσά είναι οικία αυτή η γνωμοδότηση, γιατί έχουμε ήδη εγκρίνει ένα, μια παρόμοια γνωμοδότηση πριν από δύο χρόνια, όταν η κυρία Μουνίθ ήταν η συγγήτριά μας. Και είναι αυτή η βάση για τη σημερινή μου γνωμοδότηση. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν απέτυχε αυτή η διαθεσμική διαδικασία για άσχετους λόγους. Εσείς ξέρετε, θυμόσαστε κύριε Μπροκιατή, ήταν μια από τις μεγάλες μάχες μεταξύ Κομισιών Κοινοβουλίου και Συμβουλίου η οποία παρέμεινε σοντανή μέχρι και σήμερα. Έχουμε λοιπόν δύο νέα σχέδια. Ένα για, το, για τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές και η άλλη η διαθεσμική συμφωνία για τα θέματα του προπολογισμού. Δεν έχουν αλλάξει πολλά από την εποχή αυτή. Έχω ε, συμπεριλάβει λοιπόν πολλά στοιχεία από την έκθεση της κυρία Μουνίτ που ήταν πολύ καλή και ανεκρίτη στην Επιτροπή μας. Οι δύο βασικές ιδέες να καταργήσουμε τους πυλώνες οι οποίες υπήρχαν για την ε, ΚΕΠΑ και να ενσωματωθεί πλήρω η ΚΕΠΑ στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, να αυξήσουμε και την ευκαμψία της ε, χρηματοδότησης της ΚΕΠΑ και τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτήν και δύο νέα στοιχεία. Καταρχήν εγώ ζητώ να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία από τον προπολογισμό της ΚΕΠΑ να υπάρξει ένα κεφάλαιο για την ΚΕΠΑ στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να υπάρχει ένα χωριστό κεφάλαιο για κάθε δράση της ΚΕΠΑ και για κάθε συγκεκριμένο ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν θα αυξήσει την ευκαμψία, θα μας δώσει μάλλον μεγαλύτερη ευκαμψία να μετακινούμε ποσά μεταξύ των ε, αντιπροσωπιών. Αυτό δεν θα το χάσουμε. Επίσης ζητάμε από την Κομισιόν να έχει μέσα στην ίδιο τίτλο του προϋπολογισμού να έχει ξεχωριστές γραμμές για κάθε περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιδράσει με έναν τρόπο που είναι εύκαμπτος και ταχύς, αλλά θέλουμε συγχρόνως να έχουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια για το πού πηγαίνουν τα λεφτά. Φέρνουμε πολιτική λογοδοσία χωρί να χάσουμε την ευκαμψία. Αυτό θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να θεσπίσει πολιτικέ προτεραιότητε με το να δίνει συγκεκριμένα ποσά, παραδείγματο για ειδικέ αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι το θέμα των κοινών συναντήσεων διαβουλεύσεω, όπω αναφέρονται. Εκεί πέρα πραγματοποιείται η καθημερινή παρακολούθηση των δράσεων της ΚΕΠΑ και ο στόχος μας είναι να γίνουν αυτές οι συναντήσεις πιο αποτελεσματικές με το να θέσουμε πιο ανάγλυφα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτές οι συνεδριάσεις και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών. Ζητούμε επίσης να καθοριστεί και η σύνθεση των συμμετεχόντων για να γίνει πιο αντιπροσωπευτικές αυτές οι συναντήσεις και ο στόχος μας είναι να υπάρχουν καλύτερες παροχές εκθέσεων για τις υπηρεσίες αυτές προ την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και πιστεύουμε ότι όπω και η προηγούμενη έκθεση Μουνίθ που ενεκρίθηκε το 2010 ακολουθεί το πνεύμα τη συνθήκη Λισαβόνα και θα βοηθήσει να έχουμε μεγαλύτερη πολιτική λογοδοσία και καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο στην ΚΕΠΑ με το να συγχρόνω αυξήσει την ε, ευκαμψία τη πολιτική αυτή και περιλαμβάνω και ένα χρονοδιάγραμμα <clears throat> στην γνωμοδότηση αυτή Σήμερα είναι η πρώτη εξέταση, η προθεσμή για τροπολογίε την Πέμπτη και η δεύτερη εξέταση το Σεπτέμβριο, αν θέλει ο Θεός, και θα ψηφίσουμε στην Αρμόδια Επιτροπή Προϋπολογισμών τον Οκτώβριο. Και επομένω η Επιτροπή Προπολογισμών είναι αυτή η οποία καθορίζει το χρονοδιάγραμμα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και προσβλέπω στα σχόλιά σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπραντνερ. Εγώ ανέλαβα το δύσκολο καθήκον να αντικαταστήσω τον κύριο Μπροκ, Προς το παρόν, η Ναντέτσκα Νέιτσκι έχει το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Όσον αφορά την διαθεσμική συμφωνία αυτή, η εκτίμησή μου είναι ότι οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν βασικά με την πρόταση της Επιτροπής. Όλοι θέλουμε να αναγνωρίσετε περισσότερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχεδιασμό και τον έλεγχο της εφαρμογής της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Απόψή μας ε, είναι να προτείνουμε συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Εγώ πιστεύω ότι το σχέδιο γνωμοδότησης κάνει ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν με τις δικές τους ιδέες και τροπολογίες. Ελπίζω ότι η θέση της ΑΦΕΤ θα στηριχθεί θετικά και από την Επιτροπή Προπολογισμών και ότι όταν φτάσουμε στη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και αυτοί θα συμφωνήσουν ότι ο μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος νομιμοποιεί ακόμα περισσότερο την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Ναντέστα Νέσκι. Άννα για Μέκε. Α, δεν είναι εδώ. Τότε... Η κυρία μου έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση της κυρίας Μπράτνερ χαρακτηρίζεται από συνοχή σε σχέση με τα όσα είπαμε και πέρυσι στα πλαίσια της διαθεσμικής συμφωνίας και η συνοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό για να κρατήσει το Κοινοβούλιο την δύναμή του στην υπόθεση αυτή. Είναι πολύ σημαντικές όλες οι τροπολογίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα η τροπολογία αριθμός 4, η οποία αναφέρεται στην δυνατότητα τα κονδύλια τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί να μπορούν να χρησιμοποιούνται καθ' την διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών και όχι μόνο μέχρι το έτος 1, 1 μη δηλαδή συν 3. Έπειτα ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπάρχει η συνοχή σε σχέση με τόσα έχουν γίνει τις προηγούμενες χρονιές. Η σοσιαλιστική ομάδα συμφωνεί και ελπίζουμε να διατηρηθεί η ομοφωνία που πετύχαμε και πέρυσι σε σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μονή. Δεν έχει ζητήσει κανένας άλλο το λόγο. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 12η Ιουλίου 12 το μεσημέρι. Ερχόμαστε τότε στο σημείο 18, ενδιάμεση έκθεση σε σχέση με το θετικό αποτέλεσμα του πολιτου δημοσιονομικου δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 με τη διαδικασία έγκρισης. Η κυρία Γιαννάκου είναι η Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η κατηγορία ε, του προϋπολογισμού ε, και στην προκειμένη περίπτωση του δημοσιονομικού πλαισίου η Ευρώπη στον κόσμο αποτέλεσε αντικείμενο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων υπερβολικά πολλών διορθώσεων και αλλαγών. Αυτό οφειλόταν τόσο ε, στο περιορισμένο της χρηματοδότηση όσο και στην έλλειψη ευελιξίας η οποία υπήρχε ώστε να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που προέκυπταν. Οι νέε αρμοδιότητε που εισήχθησαν από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγονται ορθώ μια συμπληρωματική χρηματοδότηση ώστε να μπορεί η Ένωση να διαδραματίζει το ρόλο του διεθνού παράγοντα που τη αρμόζει. Σαφέστατα υπάρχει μια ικανοποίηση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά στις πιστώσεις και για την κατηγορία 4 και για την αύξηση η οποία προτείνεται και ελπίζω να μην υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις εν συνεχεία στο επίπεδο του Συμβουλίου που θα μείωναν το αρχικά καλό ποσό το οποίο έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κλειδί για την επιτυχία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της κατηγορίας 4 θεωρώ ότι είναι ευελιξία, η οποία είναι πρωταρχικής σημασίας ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αντίδρασης σε απρόβλεπτες καταστάσεις και κρίσεις που δεν μπορούν να προγραμματιστούν, διατηρώντας ωστόσο τα θεσμικά κεκτημένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από των θεμάτων του προϋπολογισμού. Η απαραίτητη ευελιξία κατά την εφαρμογή της κοινή εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας δεν θα μπορούσε άλλωστε να δικαιολογήσει με οποιοδήποτε τρόπο απαλλαγή όσο αφορά στο ρόλο και στην ευθύνη της αρμόδιας αρχής για τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό το λόγο, στη γνωμοδότησή μου, απορρίπτω κάθε άλλη διάταξη που θα μπορούσε να εισαγάγει περιορισμούς της εξουσίας της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όπως παραδείγματος χάρη είναι η απαγόρευση εγγραφής πιστώσεων σε αποθεματικό που προβλέπεται από το άρθρο 11 της πρότασης συντονισμού του Συμβουλίου. Στην πρότασή μου προτείνω παράλληλα τη δημιουργία μιας κατάλληλης διαδικασίας για την αυτόματη ανακατανομή των μη χρησιμοποιουμένων κονδυλίων στο τέλος κάθε δημοσιονομικού έτους. Η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου ε, για το πρόγραμμα πρέπει να εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τη συμφωνία του Συμβουλίου επί των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των πόρων και των αποζημιώσεων που δημιουργούνται από τα χρηματοδοτικά μέσα. Ολοκληρώνοντας κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα της οικονομικής ενίσχυσης προς τις υποψήφιες να εισαχθούν χώρες και τις δυνητικά υποψήφιες χώρες, ανταποκρινόμενοι στην αρχή more for more και επιβραβεύοντας έτσι τις προσπάθειες και την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη και τις δυνατότητες υποδοχής της Ένωσης, absorption capacity. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιαννάκου. Η Άρια Μουνίθ ως πρώτη σκιώδης εισηγήτρια. Μαρία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάνει μια θετική αξιολόγηση της πρότασης Κομισιόν η κυρία Γιαννάκου σε σχέση με τις πιστώσεις που προβλέπονται για την κατηγορία 4. 70 ε, δισεκατομμύρια για όλη την γιατί όλη την περίοδο και το ίδιο ποσό που προβλέπεται για το 2013, 1.400 για το έτος 2014. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιου παίκτη για τα θέματα αυτά και ιδίως σε σχέση με τις χώρες, τις όμορες και τις τρίτες χώρες που έχουν στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως για τη Λατινική Αμερική. Πιστεύουμε ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξη η πρόταση της κυρίας Γιαννάκου σε σχέση με τα αριθμητικά ποσά. Για το 2014 προβλέπει να μην υπάρξει καμία αύξηση σε σχέση με το ποσό το οποίο προβλέπεται για το έτος 2013. Χθες εμείς είχαμε πει ότι ο προπολογισμό δεν πρέπει να θεωρείται μοναχα ένα άχθος που να το βγάλουμε από τους ώμους μας, αλλά ένα πολιτικό εργαλείο το οποίο είναι απαραίτητο για να φέρουμε σε πέρα τα πολιτικά εγχειρήματα τα οποία θεωρούμε σημαντικά. Γι' αυτό εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Θεωρούμε ότι ο γεωγραφικός χώρος δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναφέρει και τις χώρες οι οποίες είναι στρατηγική σημασία και να δώσει μια γενική εικόνα των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αναφέρουμε και τις νέους στόχους της κατηγορίας 4 μετά από τη Συνθήκη Λισαβόνας και τη δυνατότητα να προβλέπεται από τις πλευράς προϋπολογισμού η προσαρμογή της κατηγορίας 4 σε κρίσεις ή επιτακτικές ανάγκες. Θα καταθέσουμε λοιπόν τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Γιαννάκου εάν θα μπορέσει να έχει ευμενή στάση σε σχέση με τις τροπολογίες της Σοσιαλιστικής Ομάδος. Ευχαριστώ πολύ. Η Φραντσέσκα Μπραντνερ. Γενικά θα συμφωνήσουμε με τις προτάσεις της κυρίας Γιαννάκου. Αν δει κανεί τη συζήτηση στο Συμβούλιο και τις προτάσεις για μειώσεις 10%, αν μπορέσουμε να διατηρήσουμε το παρόν επίπεδο αυτό θα είναι μια μεγάλη επιτυχία, αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος μας και θα πρέπει να δώσουμε μάχη προς την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερα για να έχουμε τη δυνατότητα υποχώρησης. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι μπορούμε να ζητάμε σε αυτή τη φάση πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αποκτήσουμε. Θα πρέπει να είμαστε σκληροί στο να κρατήσουμε αυτά τα οποία έχουμε. Γενικά το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά απαιτητικό και επιθετικό και στο τέλος της διαπραγμάτευσης να μην έχει πάρει τίποτα. Το θέμα είναι να έχουμε προτάσεις τις οποίες πράγματι μπορούμε να υπερασπιστούμε, προτάσεις ρεαλιστικές και ας προσπαθήσουμε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο να ακρατήσουμε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Η Σαμπίνα έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Εμείς συμφωνούμε για τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο γίνεται η δυνατότητα να διατηρηθεί η μεγαλύτερη ευκαμψία από την πλευρά της Κομισιόν, αλλά θέλουμε συγχρόνως να διατηρήσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θέλουμε να υποσκαφθούν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το δικαίωμα για τον έλεγχο του προπολογισμού θα πρέπει να παραμείνει αναλύωτο ακόμα και αν ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη ε, σε θέματα αρχής σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα καταθέσουμε αντίστοιχες πολιτικού χαρακτήρα τροπολογίες στη γνωμοδότηση της κυρίας Γιαννάκου. Ευχαριστώ κυρία Λόζιν. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Η Κομισιόν όχι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να λάβει το λόγο, αλλά αν δεν ε, χρειάζεται, ξαναδίνω το λόγο στην κυρία Γιαννάκου. Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις που έγιναν από τις πολιτικές ομάδες και επειδή ετέθηκε το θέμα ειδικά από τη σοσιαλιστική ομάδα, βεβαίως και μπορούμε να συνεννοηθούμε ε, και να συζητήσουμε βλέποντας τις τροπολογίες που έχει διάθεση ο καθένας να υποβάλει. Θα υπάρξει καλή διάθεση και συνεννόηση με όλους τους shadow εισηγητές. Uh, Ωραία. Έχουμε κλείσει λοιπόν αυτή την συζήτηση. 12 Ιουλίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, μεσημέρι της 12 Ιουλίου. Έρχεται η κυρία Όιουλαντ και έχουμε το θέμα της προξενικής προστασίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό. Έχετε το λόγο, Χριστίνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική και πρακτική. Έχει να κάνει με την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών εκτός επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώνονταν ειδικά σε περιπτώσεις κρίσης εκτός συνόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση τώρα συνδέθηκε με την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε περιπτώσεις τέτοιων κρίσεων ή έκτακτων καταστάσεων. Πρότειναν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλέγει μία χώρα που αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Η πρόταση βρίσκεται τώρα στα δικά μας τα χέρια. Πολλοί από τους συναδέρφους και εγώ η ίδια μεταξύ άλλων αναδείξαμε περισσότερο αυτή την ιδέα του καλύτερου συντονισμού και τώρα νομίζω ότι υπάρχει μια πλειοψηφία τουλάχιστον οι συνάδελφοί που υπέβαλαν τροπολογίες βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Δηλαδή λένε αντί να επιλέξουμε μία χώρα που έχει ηγετικό ρόλο, να μπορούμε τον ρόλο αυτό να τον αναθέσουμε στις μόνιμες αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις τρίτες χώρες. Οι λόγοι είναι πολύ και διάφοροι. Από τη μια μεριά είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε πλήρως τις νομικές διατάξεις της συνθήκης μας που μας επιτρέπουν να κάνουμε κάτι τέτοιο και δεύτερον, οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα οι μικρές, δεν έχουν ευρεία προξενική κάλυψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ τώρα έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα που έχουμε σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις να τους αναθέτουμε συντονιστικό ρόλο, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την προστασία των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρχει η συμμεταχείριση αποτελεσματική και να τους δίνεται όσο γίνεται καλύτερη προξενική προστασία. Μάλιστα, κοιτάμε κάπως ακόμα πιο μακριά. Θα μπορούσε να ήταν μια καλή ε, ιδέα να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αναλάβει εκείνη κάποιες από τις προξενικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να υπονομεύσουμε βέβαια την σημασία που έχουν οι χώρες μέλη και τα προξενία τους και παρουσία, τους, παρουσία των προξενίων τους σε τρίτες χώρες. Το λέμε αυτό για πρακτικούς λόγους, ότι ίσως έτσι μπορούμε να απλοποιήσουμε κάπως τις διαδικασίες από τις οποίες πρέπει να περάσουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά έτσι μειώνουμε επίσης και τον φόρτο εργασίας για πολλές χώρες. Συγχρόνως, τελευταίο αλλά ίσως όχι και λιγότερο σημαντικό, έτσι βελτιώνουμε και την ε, προβολή της ευρωπαϊκής ηθαγένειας ως προς τις τρίτες χώρες. Αυτή είναι η εισαγωγή που είχα να κάνω. Οι συνάδελφοι νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών μπορούμε να καταλήξουμε στην ε, τελική μας τοποθέτηση και να την υιοθετήσουμε το Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε. Νάιτσκι τώρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη παρέμβαση. Η κυρία Όγιολαντ κάνει σωστές προτάσεις σε σχέση με τη γνωμοδότησή της για την προξενική προστασία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσουν τον ρόλο προστασίας των πολιτών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα αυτών που δεν εκπροσωπούνται στη συγκεκριμένη χώρα. Και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ακολουθεί την ίδια γραμμή με τη δική μας. Κατανοώ βέβαια τις αντιρρήσεις ορισμένων συναδέλφων των ιδιαίτερα των Βρετανών αλλά παρόλα αυτά η συνθήκη έχει υποχρεώσεις ε, οι οποίες προέρχονται από τη συνθήκη και πρέπει να τη σεβαστεί και το να μην εμπλέξει κανείς τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προβλέψεις για την προξενική προστασία είναι κάτι το οποίο θεωρηθεί απαράδεκτο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να χρησιμοποιήσουν ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες των αντιπροσωπιών. Αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι η κυριαρχία των κρατών μελών αλλά η ασφάλεια των πολιτών τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για μια πραγματικά γνωμοδότηση η οποία είναι ιδιαίτερα θετική. Αυτό το θέμα το είχαμε συζητήσει και είχαμε προσπαθήσει να αντιμετωπίσουμε στην περίπτωση της δημιουργίας της υπηρεσίας εξωτερικών ε, υποθέσεων έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη προστασία ε, ε, των, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας απογοητεύει γιατί περιορίζεται στη βελτίωση του συντονισμού αλλά δεν αναφέρεται καθόλου στο ρόλο των αντιπροσωπιών. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε συνέργειες και να μειώσουμε το κόστος χωρίς ε, να δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι όταν δημιουργούνται ε, δύσκολες καταστάσεις, τα κράτη-μέλη έτσι και αλλιώς καλούνται να συνεννοηθούν. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών μας. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν είναι εμείς να ορίσουμε έναν υπεύθυνο συντονισμού στις αντιπροσωπείες. Αυτό είναι κάτι το βασικό για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορέσουμε να κάνουμε και περισσότερα βήματα, τότε θα πρέπει να αναλάβουν οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και προξενικό ρόλο, εφόσον βέβαια οι χώρες μέλη δεν θέλουν να τον έχουν αυτό το ρόλο. Υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένες χώρες, οι Βρετανοί δημιουργούν επιπλέον προβλήματα Νομίζω ότι αν δει το Ηνωμένο Βασίλειο το πόσα χρήματα μπορεί να ε, εξοικονομήσει θα αλλάξει την άποψή του. Νομίζω λοιπόν ότι σε συνεννόηση και με την κυρία Μπάουερ της Λίμπε μπορούμε να επιμείνουμε και να δείξουμε το όφελος το συγκεκριμένο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια τέτοια ρύθμιση. Συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά είχα μια κλίση από Υπουργό Εξωτερικών. Η κυρία Βερζιά που έχει δει το λόγο δεν είναι εδώ. Η προθεσμία... Α. Α, είναι εδώ η κυρία Μπάουερ. Ή όχι. Η Εντίτ Μπάουερ από την Λίμπε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίδεται. Θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Να πω ότι εκτιμώ την στάση της σχετικά με τις τροπολογίες θα ήθελα να ζητήσω να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν δύο τύποι εν πάση περιπτώσει προξενικής ε, ε, προστασίας, οι καθημερινές υπηρεσίες και η διαχείριση κινδύνων γενικότερα. Σχετικά λοιπόν με τις καθημερινές υπηρεσίες, πράγματι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν είναι η κατάλληλη για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις καθημερινές ανάγκες της προξενικές των πολιτών. Σαν παράδειγμα απώλεια διαβατηρίου κτλ. Και αν λάβουμε υπόψη μας και το άρθρο 23 της Συνθήκης της Λισαβόνας, λέγεται εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την δυνατότητα να στραφεί σε ε, εκπρόσωπο ιουδήποτε κράτους μέλους για την ανάληψη του ρόλου αυτού των προξενικών υπηρεσιών. Θα ήθελα λοιπόν να εμείνουμε, να ζητήσω να εμείνουμε στο άρθρο 23 για τις καθημερινές προξενικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο όχι. 13 Ιουνίου η προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών. Φτάνουμε τώρα στην έκθεση του Τσάρλ Στάνοκ, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κέρας. Ευχαριστώ. Μόλις ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου μου είπε ότι είναι το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε λάθος έχουμε βάλει τον τίτλο από ό,τι φαίνεται. Το Συμβούλιο πάντως έχει δημοσιεύσει τα συμπεράσματά του για το κέρα τη Αφρικής στι 14 Νοεμβρίου που μας πέρασε, οπότε η έκθεσή μου αποτελεί μια ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιδράσει και να διευκρινίσει. Στρατηγικό πλαίσιο για τη διακυβερνητική αρχή όπου συμπεριλαμβάνονται 8 χώρες. Το πώς ορίζει κανείς το κέρας της Αφρικής ε, βέβαια εξαρτάται είναι η Ερυθρέα, αν και ε, εξαιτία ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει φύγει, και Ένια, Σομαλία, Σουδάν, Ουγάντα και Νότιο Σουδάν. Είναι μια περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη αστάθεια. Δεν υπάρχει πολιτική ούτε οικονομική σταθερότητα. Αυτό είναι γνωστό σε όλους μας όσον αφορά την Σομαλία. Υπάρχει το Σουδάν με τον Νότιο Σουδάν που βρίσκονται σε διένεξη. Υπάρχει ανάμεσα στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα επίσης ένταση και ανάμεσα και στην Ερυθρέα και το Τζιμπούτι. Οπότε τελικά το κέρας της Αφρικής δείχνει να είναι η πιο επικίνδυνη περιοχή στον κόσμο. Πάντως υπερβάλλουμε όσον αφορά την αστάθεια, επειδή υπάρχουν ε, και άλλοι παράγοντες. Υπάρχει η πείνα, υπάρχει η πειρατεία, υπάρχει η διακίνηση ναρκωτικών, και όχι μόνο και άλλων ε, παράνομων προϊόντων, ε, ενισχύονται τρομοκρατικές ομάδες εκεί. Αυτοί είναι κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μας οδηγούν στα συμπεράσματα αυτά. Μιλάει για στρατηγική στην περιοχή το Συμβούλιο να υπάρχει μια στρατηγική βάση της οποίας ε, να λογοδοτεί το Συμβούλιο και να μπορούμε να διορθώσουμε κάπως την κατάσταση. Η ασφάλεια στην περιοχή να είναι τέτοια από την οποία να μην κινδυνεύουν ε, οι γείτονες ε, χώρες, μείωση της ένδειας και στήριξη της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας επιτόπου. Εδώ επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω κάποιους τομείς. Η Σομαλία, για παράδειγμα, σίγουρα είναι πολύ κρίσιμη στιγμή που ζει η χώρα. Γιατί εδώ και δεκαετίες υπάρχει αστάθεια και η εντολή της μεταβατικής κυβέρνησης εκπνέει τον, Οκτώβριο, το, συγγνώμη, τον Αύγουστο που μας έρχεται, τον επόμενο μήνα δηλαδή. Άρα χρειάζεται πολιτικός διάλογος και να στηρίξουμε την οργάνωση ελεύθερων εκλογών εκεί. Επίσης πρέπει να υπάρξει συνένεση για να στηριχθεί η νέα κυβέρνηση της Σομαλίας. Η προθεσμία για τροπολογίες είναι η 8 Σεπτεμβρίου στην έκθεσή μου, δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές στην Σομαλία, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν και την άποψή τους για τις εκλογές εκεί. Άλλο θέμα, όπως είπαμε, είναι η πειρατεία, η οποία βέβαια και κοστίζει πάρα πολύ στο διεθνές ε, εμπόριο μέσω ναυτιλίας. Έπειτα υπάρχει το θέμα των όπλων. Χρειάζονται τροποποίησεις για να υπάρχει έλεγχος όσον αφορά τα όπλα στην πολεμική βιομηχανία, πράγματα τα οποία προς το παρόν βέβαια κοστίζουν πάρα πολύ. Πάντως θα υποβάλω τροπολογίες για τα ζητήματα αυτά. Να μην ε, χειροτερεύει η ανασφάλεια στην περιοχή εξαιτία της πειρατείας. Υπάρχει Αταλάντα όπου προτείνονται ε, διάφορα πράγματα κατά της πειρατείας. Ίσως γνωρίζετε ότι 20 Μαρτίου το Συμβούλιο παρέτεινε την, αποστολή, την εντολή δηλαδή της αποστολής Αταλάντα μέχρι το 2014 ώστε να μπορέσει να συμπεριλάβει και την πειρατεία on Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε στον τομέα της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας και να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές, όπως για παράδειγμα απασχόληση γενικότερα στη Σομαλία. Θα ζητάω επίσης και δικαιοσύνη σε διάφορα συστήματα της χώρας να συλλαμβάνονται οι πειρατές και να υπάρχει δυνατότητα της δικαιοσύνης μέσω υποδομών για να υπάρχουν φυλακές, ε, οι πειρατές που καταδικάζονται να μπαίνουν στη φυλακή κτλ. Αυτές οι περιοχές δηλαδή και αυτές οι χώρες να μπορούν να συλλαμβάνουν και να φυλακίζουν τους πειρατές. Υπάρχει πρωτοβουλία για να ενισχυθεί βέβαια και η ναυτιλία και η δικαιοσύνη, εκπαιδεύοντας και βοηθώντας τους φύλακες. Υπάρχουν τώρα και άλλοι διεθνείς εταίροι, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν όσον αφορά την αυτιλία. Στην έκθεσή μου λοιπόν μιλάω ιδιαίτερα για την Αθιοπία, την Κένια που δίνει στρατό στην Άμασον, του Ουγκάντα όπου εκπαιδεύονται ευρωπαϊκές δυνάμεις για να βοηθήσουν στη σταθερότητα. Η διεθνής κοινότητα τώρα Πρέπει να δούμε τι προσπάθειες κάνει. Το βέβαιο είναι ότι η Αφρική πρέπει να αποφασίσει και να δράσει από μόνη της. Γι' αυτό μιλάω για την Αφρικανική Ένωση και για την διακυβερνητική αυτή ένωση, την ΕΚΑΤ που σας είπα πριν. Έχουμε και άλλα παραδείγματα στο κέρας της Αφρικής. Μια ΖΙΕΤ που δεν αναγνωρίζεται. Μιλάμε για την Σομαλιλάνδη είναι ένα θετικό παράδειγμα που κατέδειξε την ικανότητα για ανάπτυξη και δρέωση δημοκρατικών, οικονομικών και διοικητικών δομών. Συνεργαζόμενοι με τη διεθνή κοινότητα για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και της πειρατείας. Τέλος αναφέρομαι και σε άλλες περιοχές όπου πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει λύση και που υπάρχουν εντάσεις για να αποφύγουμε εντάσεις και στο μέλλον. Για παράδειγμα, επήγει να υπάρξει μια συμφωνία ώστε να μοιραστούν τους φυσικούς τους πόρους του Σουδάν με τον Νότιο Σουδάν και να μην υπάρξει άλλη διένεξη μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Να μπορέσει να γίνει βιώσιμο το Νότιο Σουδάν που είναι μια χώρα που πρόσφατα φτιάχτηκε. Περιμένω τα σχόλιά σας αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη σήμερα. Σα είπα, 8 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών, 10 Οκτωβρίου για να ψηφίσουμε και τον Νοέμβριο στην μήνυ σύνοδο στις Βρυξέλλες θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ Τσάρλς. Ήδη ανακοίνωσε στην προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών που είναι κανονικά ευθύνη του Προέδρου και θα το κάνω έτσι και αλλιώς στο τέλος της συζήτησης. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Συζήτησα με τον σκιώδη συγητή του ΕΛΚ που δεν μπορεί να είναι παρόν και μου ζήτησε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Δεν ήξερα ότι θα είμαι εδώ του Προέδρου, αλλά αυτό δεν θα με εμποδίσει. Ελπίζω να κάνω τις παρατηρήσεις αυτές. Ο κ. Βένσον θέλει να ευχαριστήσει τον κύριο Τάνοκ το κέρας της Αφρικής είναι μια περίπλοκη περιοχή, οι προκλήσεις είναι τεράστιες και γι' αυτό οι στρατηγικές και οι αναλύσεις απαιτούν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο κύριος Σβένσον θα μελετήσει την πρόταση του κύριου Τάνοκ προσεκτικά και θα καταθέσει επικοδομητικές τροπολογίες. Η πρόταση του κύριου Τάνοκ, η αρχική, είναι μια καλή ε, αρχή, αλλά ο κύριος Βένσον θα ήθελε να εμείνουμε περισσότερο σε ορισμένες πλευρές. Η κατάσταση θα πρέπει να συγκεντρώσει την η εξέταση θα πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί η κατάσταση εκεί είναι πάρα πολύ κακή. Το δικαίωμα στη ζωή, στην ασφάλεια, στην υγεία είναι το μεγαλύτερο δεοντολογικό δίλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον κόσμο και γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστεί με τους πρωταγωνιστές της περιοχής, με τις κυβερνήσεις της περιοχής για να δοθούν εγγυήσει. Και τα δικαιώματα των γυναικών επίσης έχουν αγνοηθεί επί μακρόν ο φανατικός Ισλαμισμός έχει επίσης επεκταθεί στην περιοχή και αυτό δημιουργεί προβλήματα και κινδύνους στις θρησκευτικέ μειονότητες. Υποστηρίζοντας την ασφάλεια στην περιοχή θα διασφαλίσουμε και την καταπολέμηση της πειρατείας και τις παράνομες δραστηριότητες και ε, γενικότερα να δώσουμε την δυνατότητα στην οικονομία και στο εμπόριο να αναπτυχθούν. Παραδείγματα καλύτερης διακυβέρνησης έχουμε όπως το Σομάλιλαντ και θα πρέπει να υπογραμμιστούν σαν πρότυπο θα έλεγα και για άλλα μέρη της Σομαλίας. Και ο κύριος Βένσον τελειώνει λέγοντας ότι καλή τύχη στον κύριο Τάνοκ με αυτό το εξαιρετικό ψήφισμα. Έπρεπε να σας μεταφέρω λοιπόν το μήνυμα αυτό. Η κυρία Μουνίζη έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Τάνοκ για την, ε, το σχέδιο έκθεσής του. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή βάση να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά και θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε με διάφορες πτυχές που για μας η σοσιαλιστική ομάδα μας φαίνεται ότι ελείπουν από την ε, έκθεση του κυρίου Τάνοκ. Καταρχήν θέλαμε να αναφέρουμε πιο πολύ σε βάθος την ανθρωπιστική κρίση και την ιδέα της πρόσβασης στους ανθρώπους του ίδιους Υπάρχει κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για οποιαδήποτε έκθεση για το κέρας της Αφρικής. Δεν υπάρχει αναφορά για αυτές τις μετακινήσεις, για τη διασπορά της περιοχής αυτής, ε, του ομαλού δηλαδή και τους άλλους που βρίσκονται στη διασπορά. Και επίσης θεωρούμε <clears throat> ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η διάσταση του φύλου σε όλα τα στάδια της επίλυσης αυτής της σύγκρουσης και επίσης η αποστράτευση και η των ε, μαχητών είναι απαραίτητη για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη, το οποίο θα επιτρέψει να επανέλθουμε σε δράσεις ανάπτυξης. Ούτε αναφέρεται η ανάγκη να επιτευχθούν τις ανάπτυξη τη χιλιετία, να μειωθεί η πείνα και η ένδια και να χρησιμοποιηθούν οι ανανεώσιμοι πόροι για την ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να αναφερθούν σε μια τέτοια έκθεση. Είναι πτυχές λοιπόν που είναι νευραλυγικές για αυτή την περιοχή και πρέπει να κατανοήσουμε ότι συνδέονται ε, απόλυτα μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε τα θέματα της ανάπτυξης με τα πολιτικά θέματα. Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μια αποσταθεροποίηση της περιοχής υπάρχει μια μεγάλη αστάθεια και επίσης και οι σχέσεις σταθερότητος και ανάπτυξης περνά και μέσα από την αντιμετώπιση της κλιματικής ε, αλλαγής. Είναι πάρα πολλοί τρωτοί αυτοί οι οποίοι έχουν τύχει εσωτερικού εκτοπισμού και οι πρόσφυγες. Σε σχέση με την πειρατεία αναφέρει τις δύο απόστολες Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Στάνοκ, την Ευρωαφόρ και την ε, Αταλάντα και υπάρχει και η επόμενη ε, αποστολή Eurocup Nestor. Εγώ σύμφωνο απόλυτα για τα θέματα αυτά που αναφέρει, αλλά και πάλι από την οπτική γωνία της σοσιαλιστικής ομάδας θα πρέπει να αναφέρουμε την ανάγκη να υπάρξει και κάποιος έλεγχος για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν φρουρούς για τον Ινδικό ωκεανό. Χρειαζόμαστε ένα οδικό χάρτη και κάποια πρότυπα για να καθοριστούν καλύτερα οι ευθύνε του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να υπάρξει ένα κώδικα συμπεριφορά και αυτό είναι μια ευκαιρία να ζητήσουμε από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να αναλάβουν μια πρωτοβουλία στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με τον εισηγητή και τι άλλε πολιτικέ ομάδε για αυτή την τόσο σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μουνίθ. Ο Ράινερ Μπουτικόφ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για το σχέδιο που έχει ετοιμάσει και που μας παρουσίασε σήμερα. Όπως και αυτός, έτσι και εγώ σκοπεύω να παίξω επικοδομητικό ρόλο. Πιστεύω όμως ότι μας μένει αρκετή δουλειά. Μια βασική αρχή που υπογράμμισε ο εισηγητής και με την οποία είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να απορρέει από την Αφρική. Είναι αφρικανική υπόθεση και η Αφρική πρέπει να έχει τον ηγετικό ρόλο. Θέλω πάντως να υπογραμμίσω πέντε σημεία κάπως σύντομα, στο οποίο έχω κάπως διαφορετική άποψη. Πρώτον, για τις ε, γείτονες χώρες. Είμαι πιο επικριτικό όσον αφορά τον ρόλο που χώρες όπως η Αιθιοπία έχουν παίξει με τις μονομερείς τους δράσεις. Και ίσως θα έπρεπε να αναφέρουμε εδώ και το γεγονός ότι η Ερυθρέα έχει κατηγορηθεί από την ε, ομάδα του ΟΗΕ ε, τη στηρίζει τον Αλσαμπά. Είναι δηλαδή μια αρνητική και αυτή συμπεριφορά. Δεύτερον, Μιλάμε για το στρατηγικό πλαίσιο όσον αφορά το κέρας της Αφρικής. Όμως, εδώ μπερδεύονται πολλά πράγματα. Μια αλλαγή που θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά είναι εάν ο ειδικό απεσταλμένος ο Αλεξάνδρ Ρότος εάν θα μπορούσε να έχει ηγετικό ρόλο συνολικά για το θέμα ίσως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να ενισχύσουμε το ρόλο του. Τρίτον, εγώ κρίνω κάπως πιο επικριτικά της, ε, τη στρατιωτική ανάπτυξη και τις εξελίξεις εκεί. Η πειρατεία, αν έχει ανέβει παραπάνω, οφείλεται μάλλον στο Μανσούν παρά σε στρατιωτική στρατηγική που ακολουθήσαμε εμείς. Αν δηλαδή έχει μειωθεί κάπως η πυρετή και το τελευταίο καιρό. Στη συνέχεια, είμαι πολύ επιφυλακτικός να δω πώς προτείνει τελικά να αντιμετωπίσει το θέμα της ανεξαρτησίας της Σομαλιλάνδης ο εισηγητής ζητάει να αναγνωριστεί σαν ε, χώρα, ανεξάρτητη. Είναι πολύ λεπτό όπως καταλαβαίνετε. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να υπογραμμίσουμε τη θετική συνεισφορά της Σομαλιλάνδης υπέρ της σταθερότητας στην περιοχή, αλλά δεν θα ήθελα να ενθαρρύνουμε κινήσεις ε, ανεξαρτησίας. Και θα ήθελα να τονίσουμε περισσότερο τη συνταγματική διαδικασία η οποία λαμβάνει η χώρα επί του παρόντος. Νομίζω ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος και δεν θα έπρεπε να διστάσουμε να το στηρίξουμε αυτό. Ευχαριστώ. vielen Dank. Ευχαριστώ κύριε Μπιτικόφερ. Η κυρία Λέζιν έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του, αλλά θα έπρεπε να πω από εξ αρχής ότι από τη δική μας πλευρά υπάρχουν πολλές διαφορετικές οπτικές με, την, ε, το περιεχόμενο της έκθεσης του κυρίου Τάνοκ. Συμφωνώ με τον κύριο Μπιτικόφερ και με άλλους ομιλητές ότι πρέπει να σκεφτούμε και τους ανθρώπους στην Αφρική και να τους δώσουμε τη δυνατότητα αυτή να συμμετάσχουν στην επίλυση του προβλήματος δεν πρέπει όμως να χάσουμε και από τα μάτια μας τις αιτίες αυτού του προβλήματος και τις επιπτώσεις του. Τα προβλήματα λοιπόν των, ε, της ένδυας στην περιοχή αυτή, η, η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και της Ινδίας και της Κίνας για την υπερεαλίευση στα νερά αυτά του κέρατος της Αφρικής δεν αναφέρεται πουθενά. Ο εισηγητής επίσης αναφέρθηκε στην ένδια στην αρχή, αλλά η έκθεσή του δεν περιέχει περίπου τίποτα σε σχέση με το πρόβλημα της ένδια στην περιοχή αυτή, γιατί αυτή είναι και μία από τις κύριες αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στο κέρας της Αφρικής και έχει μία πάρα πολύ αρνητική, ε, υπάρχει μία πάρα πολύ ε, αρνητική στάση των βιομηχανικών κρατών που είναι η αιτία αυτής της ε, ένδυας στην Σομαλία και σε άλλες χώρες. Αυτό πρέπει να επικριθεί και πρέπει να αναφερθεί στην έκθεση ο ρόλος λοιπόν, των βιομηχανικών χωρών. Αναφέρεται επίσης και για άλλες χώρες όπως είναι η Κένια, η Ουγγάντα και η Αιθιοπία αλλά αναφέρεται μόνο σε αυτές οι οποίες συμφωνούν με την τωρινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε με το κέντρο της Αφρικής. Δεν αναφέρεται όμως η έκθεση αυτή καμία πρόταση για να μπορέσουν να σταματήσουν οι εμφύλιες σειράξεις στην Σομαλία. Οι στρατιωτικές πτυχές του προβλήματος νομίζω ότι αντιμετωπίζονται σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο και υπερθεματίζει ο εισηγητής σε σχέση με τις στρατιωτικές αυτές ε, πτυχές, η υποστήριξη της εκπαίδευσης των ακτοφυλακών κτλ. Εμείς θα πρέπει να συζητήσουμε σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν σε μια τέτοια α, ε, στην περίπτωση της Σομαλίας να έχουμε μια δική μας εκθέση. Εμείς θα καταθέσουμε πάντως τροπολογίες προς την εκθέση του κυρίου Τάνοκ. Ο Τσάρλς θέλετε να κλείσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία τα σχόλια τα οποία έχετε μεταφέρει από τον κύριο Σφένσον, εγώ τα χαιρετίζω ιδιαίτερα. Αυτή είναι μια έκθεση η οποία αναφέρεται ιδίω στα θέματα πολιτικής Εξωτερική πολιτική και ασφάλεια ανέφερα τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρί περαιτέρω έμφαση. Θα χαιρέτησα και τροπολογίες προ την κατεύθυνση αυτή, ιδίω όταν επικαλύπτονται με τα σχόλια της κυρίας ε, Μινιούς σε σχέση με τα άτομα που είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Σίγουρα είναι προβλήματα, πρόβλημα τόσο περιοχέ που ελέγχει η Al-Shabaab και επομένως θα υποστήριζα τις τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν έχω αρκετό χώρο στη γνωμοδότηση υπομορφή χαρακτήρων, αριθμού χαρακτήρων και γι' αυτό απολογούμε. Για το θέμα το οποίο ανέφερε η κυρία Μουνίθ, συμφωνώ με την ανάγκη να αφοπλιστούν και να αποστρατευθούν οι πολιτοφυλακές, αλλά τις λέω και πάλι δεν είναι μία έκθεση Επιτροπής ε, Ανάπτυξης Επιτροπής Περιβάλλοντος. Επομένως δεν αναφέρομαι στους στόχους της χιλιετίας ή στους, ε, στην κλιματική αλλαγή γιατί δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη γνωμοδότηση και πάλι χαιρετίζω τις ε, τροπολογίες. Εγώ υποστηρίζω το να υπάρχουν ενόπλοι φρουροί στα πλοία που διέρχονται από την περιοχή αυτή γιατί δεν έχει ακόμα υπάρξει επιτυχής πειρατεία σε ένα πλοίο που έχει ένοπλη φρουρά και πάλι εγώ θα υποστηρίξω με τροπολογίε αυτή την άποψη και περιμένω να δω τι έχουν να πούν και άλλε ομάδε. Ο κύριο Κόφερ, εν συντομία, αναφέρθηκε στην ε, ε παρέμβαση άλλων χωρών όπω είναι η Αιθιοπία. Η Αιθιοπία είναι μια πηγή σταθερότητα. εν μέρη, αλλά δεν είναι απόλυτα δημοκρατική χώρα και έχει προβλήματα στο εσωτερικό της, όχι τόσο άσχημα όπως η Ερυθρέα, αλλά κάποτε θα πρέπει να δράσει και προς το συμφέρον το δικό του και να αντιμετωπίσει την επεκτατική στάση της Άλσου Shabaab στο κέρας της Αφρικής. Ανέφερα στο ότι θα πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη ε, διατύπωση αναφερθήκατε στο ότι σε εποχή μουσόνος η πειρατεία μειώνεται, αλλά η πειρατεία ήδη μειώθηκε το 2011, αυτό το δείχνουν και οι στατιστικές που είδαμε από την αποστολή Αταλάντα. Πιστεύουμε ότι η πειρατεία έχει μειωθεί σημαντικά, έχει μειωθεί πάρα πολύ η ικανότητα των πειρατών να προβαίνουν αποτελεσματικές ενέργειες, παρά όλα αυτά πρέπει να διατηρηθεί η πίεση και υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η κυρία Λέζινγκ θεωρεί ότι όλα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ε, ένδυας. Διαφωνώ μαζί της, είναι ένας, ε, ε, ένας ρόλος, ένας, παίζει κάποιο ρόλο. Αλλά δεν υπάρχει καθόλου πειρατεία η οποία εκπορεύεται από την Σομαλιλάνδη, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ φτωχή. Επομένως δεν είναι η ένδια που τα προξενεί όλα. Δεν είναι ο μόνος λοιπόν λόγος της πειρατείας η Ένδια, γιατί θα υπήρχε σε όλη την περιοχή της Σομαλίας. Η Σομαλιλάνδη έχει καλή διακυβέρνηση, έχει δημοκρατία, έχει κάτω δικαίου. Επομένως πρέπει να διαφωνήσω με την κυρία Λόζιν για το θέμα των αιτιών της πειρατείας για τη Σομαλιλάνδη. Εγώ θα ήθελα να έχω μια πιο ισχυρή υποστήριξη. Εγώ υποστηρίζω την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης και την, και την αναγνώρισή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, παρέμειναν μέσα στα πλαίσια της ε, Σομαλίας μέχρι το 1991 είναι πολύ πιο ισχυρή η επιχειρηματολογία για την ε, ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης από την παραγματικά για το Κοσφοπέδιο. Εγώ δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες προτιμώ να έχω μια ουδέτερη θέση παρά να προωθήσω τη δική μου άποψη για την ανεξαρτησία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όμως το γεγονός ότι είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα της Σομαλιλάνδης. Δεν είπε κανείς κάτι υπέρ κατά της ανεξαρτησίας. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί εσωτερικά μεταξύ της Σομαλίας και της Σομαλιλάνδης. Ξέρω θα είναι ένα δύσκολο θέμα όπως μπορείτε και εσείς να φανταστείτε. Πρέπει όμως να αναγνωρίσετε ότι υπάρχουν πολλές θετικές πτυχές της Σομαλιλάνδης, της λειτουργίας Σομαλιλάνδης, αυτό που προσπαθώ να κάνω στην οικία παράγραφο και ανέφερα προς την κυρία Λέζιν ότι θα είμαι έτοιμο να δω και το θέμα της λειψιδρίας στην περιοχή της, ε, του κέρατος της Αφρικής, αλλά αυτό είναι και ένα συνολικότερο θέμα και επίσης το θέμα της υπεραλίευσης από την Κίνα και την ε, Ινδία είναι σημαντικό θέμα, όπως και η υπεραλίευση από ισπανικά σκάφη. Αλλά τα θέματα δεν είναι μοναχά οικονομικά, έχουν να κάνουν και με οργανωμένο έγκλημα, έλλειψη κράτους δικαίου, ε, έλλειψη ελέγχου, το γεγονό ότι είναι ένα αποτυχημένο κράτο η Σομαλία. Αλλά εγώ είμαι έτοιμο να συζητήσω τι τροπολογίε με όλου του κοιόδου εισηγητέ για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιε συμβαστικέ θέσει. Σα ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο Πέτρινγκ. 18 Σεπτεμβρίου είναι η πρόθεσμη για τι τροπολογίε του 2012 το μεσημέρι. 18 Σεπτεμβρίου θα ξανασυνεδριάσουμε στις 3 η ώρα για να ακούσουμε την Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, την Δόκτωρα Ερατό Κοζάκο Μαρκουλή και σας εύχομαι καλή όρεξη εάν θα φάτε το μεσημέρι.